καθιστούν τις κυρίες Νάιτ Σότεμπρουκ και τον κύριο Λουίς Ιντε αντιστοίχως. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού για τις ευρωεκλογέ και το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού του Κοινοβουλίου καλωσορίζω τις ε, συναδέλφους οι οποίες βεβαίως θα συμμετέχουν πλήρως με όλα τα δικαιώματα στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου υπό την προϋπόθεση πως έχουν δηλώσει γραπτός πως δεν κατέχουν κάποιο αξίωμα το οποίο είναι ασυμβίβαστο με αυτό του Ευρωβουλευτή.